Good afternoon, ladies and gentlemen. I think it's time we started. Nine minutes into our schedule. We have a very, very important... Ξεκινάμε με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Στα αριστερά μου κάθεται ένα, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ με μεγάλη χαρά Καλωσορίζω το φίλο μας, τον Επίτροπο κύριο Πίλμπαξ, για να μας μιλήσει για την τρέχουσα ε, κατάσταση του προγραμματισμού του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Όπως γνωρίζουμε, η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεαστεί από σημαντικούς παράγοντες ε, στο μέλλον. Το 2013 τελειώνει η τρέχουσα δημοσιονομική προοπτική και εξετάζουμε το DCI και το European Development Fund, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Δύο από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους στον κόσμο, λήγουν περίπου την ίδια εποχή. Είδαμε την πρόταση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που δημοσιεύτηκε από την Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα και εξ ονόματος όλης της Επιτροπής ε, επικροτούμε τις ε, σημαντικές αυξήσεις που προτείνει η Κομισιόν ε, σε εποχές οικονομικών περιορισμών. Τόσο για το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, όσο και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. θέλουμε να επιτυγχάνεται 0,7 του ΑΕ. Η ίδια πρόταση περιλαμβάνει μια δέσμευση βελτίωσης ε, της, ε, του δημοκρατικού ελέγχου των δαπανών, των χρημάτων των φορολογουμένων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατεξουσιοδότησης πράξεων. Η κατεξουσιοδότηση πράξης ε, ε, είναι κάτι το που έχουμε συζητήσει με την Κομισιόν και προσβλέπουμε στο να λάβουμε μια πιο λεπτομερή απάντηση της Κομισιόν ε, για αυτό το θέμα. Χωρίς λοιπόν άλλη καθυστέρηση, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας δίνω το λόγο με αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη εισαγωγή και παρουσίαση και είναι μεγάλη μου τιμή που έρχομαι να μιλήσω εδώ σε αυτή την Επιτροπή είναι μεγάλη ευθύνη και ευχαριστώ για την ευγένεια σας. Παίρνω τη δουλειά μου πάρα πολύ σοβαρά γιατί είμαι υπόλογος και στις αρχές του προϋπολογισμού. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε. Είναι αλήθεια ότι πρόσφατα επισκέφθηκα και όλες πολλές ε, χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Τζιμπουτί και το Σεντ Κίτσεν Nevis, ε, σε όλα αυτά τα μέρη πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πως ε, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαστε υπερβολικά χαμηλών τόνων για το τι έχουμε επιτύχει σε αυτές τις ε, περιοχές. Έχουν γίνει πολλές. Πρέπει να είμαστε επικριτικοί, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Μας συγχαίρουν για πράγματα που έχουμε Επιτυχεί, αλλά να προσπαθούμε, πρέπει να προσπαθούμε να μάθουμε και να αποκομίζουμε τα μαθήματα. Να βλέπουμε πού ήμασταν επιτυχείς και πού λιγότερο. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικά ζητήματα. Ζητήματα πολιτικής ε, και οικονομικά ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα σχετίζονται μεταξύ τους καθώς μιλάμε για ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στο πλαίσιο του οποίου ε, προσπαθούμε να επισημάνουμε τις προτεραιότητες, ε, τα αποτελέσματα. Έτσι προσπαθούμε να επιτύχουμε το στόχο της ε, ενημερωμένης αναπτυξιακής πολιτικής μας. Έχουμε ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις εντός της Επιτροπής. Το σχετικό έγγραφο θα υποβληθεί σε αυτή την Επιτροπή, θα παρουσιαστεί σε αυτή την Επιτροπή. Οι προοπτικές για τις εργασίες μας είναι πολύ καλές λόγω πρώτα απ' όλα της τρέχουσας κατάστασης της πολιτικής θα ξεκινήσω ε, λέγοντας ε, μελετώντας λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής μας ότι Είχαμε την ε, εκτενή έκθεση του κυρίου Κάτσμαρεκ και χαίρομαι που βλέπω ότι όταν μιλάμε για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ε, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Οι απόψεις μας είναι οι ίδιες για τα περισσότερα μείζωνα ζητήματα. Αναπτυξιακή πολιτική σημαντικών αποτελεσμάτων, διακυβέρνηση, ανάπτυξη των ανθρώπων είναι μερικές από τις πτυχές. Είμαι πεπισμένος ότι η πρόταση που θα προσφέρουμε το πορό θα γίνει αποδεκτή. Θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρνς για την πολύτιμη συμμετοχή του σε μια άλλη πολύ σημαντική πολιτική συζήτηση που αφορά την υποστήριξη του προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα. Ε, ακούστηκαν ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα, την αξία της επένδυσης και γενικότερα ζητήθηκε από την Κομισιόν να προβεί σε περαιτέρω βελτιώσεις ε, της ε, υποστήριξης προϋπολογισμού και σήμερα ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις για την εκθέση που θα σας παρουσιαστεί και όλα αυτά συμφωνούν με την εκθέση του κυρίου Γκέρενς. Υπάρχουν πολύ σαφείς αλλαγές οι οποίες προτείνεται να γίνουν για το ε, δημοσιονομική στήριξη στο μέλλον, εφόσον εγκριθεί. Έχουμε λοιπόν κοινέ απόψεις οι με οι οποίες με κάνουν και ελπίζω ότι θα μας εμφανιστούν καινούργιες ιδέες καθώς θα προχωράμε, οι οποίες θα έχουν την υποστήριξη της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την αναπτυξιακή χρηματοδότηση, υπάρχει μια πρόταση αύξηση της χρηματοδότησης για την εξωτερική δράση, η οποία θα βοηθήσει τις κυριότερες προτεραιότητές μας. Στο επίπεδο χρηματοδότηση που προτείνεται, ε, αποτελεί αναγνώριση των στρατηγικών στόχων που στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης και των διεθνών απαιτήσεων καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφιερώσει το 0,7 του ακαθάριστου εγχωρίου εισοδήματος ε, στην ανάπτυξη, στην υποστήριξη της ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει το μεριδιό της στις κοινέ προσπάθειες ε, χάρη σε αυτή τη στήριξη θα, δείξουν, θα δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αποφασιστικότητά της να βοηθήσει τους στοχότερους στον κόσμο. Έτσι θα έχει λάβει ένα αποφασιστικό βήμα για την επίτευξη των ε, ε, αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ωστόσο, η επιτυχία των προσπαθειών, των αναπτυξιακών προσπαθειών μας δεν εξαρτάται μόνο από τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να βρούμε τις σωστές δομές για τη χρηματοδότηση. Από άποψη δομών δεν θελήσαμε να επανασχεδιάσουμε τα πάντα. Θεωρήσαμε ότι χρειάζεται απλά να απλοποιήσουμε και να επικεντρωθούμε στα τρέχοντα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις. Θα εστιαστώ εδώ σε δύο θεμέλιους ε, λίθους ε, της αναπτυξιακής χρηματοδότησής μας που θα λάβουν ε, μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού στο νέο πλαίσιο. Θα ξεκινήσω με το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης προτείνει την ε, εκχώρηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ για τις ε, χώρες ΑΚΕ. Μιλάμε για 321 εκατομμύρια ευρώ για τα OCT. Αυτό αποτελεί ένδειξη της συνεργασίας μας ε, ενώπιον των εταίρων μας. Η Κομισιόν πρότεινε να ενταχθεί το EDF ε, στον προϋπολογισμό. Βάσει της συμφωνίας του Κοτονού, οι συνθήκες για αυτό δεν πληρούνται ακόμη απόλυτα. Ωστόσο, η προοπτική μελλοντική ένταξη είναι ρεαλιστική. και θέλουμε να εντάξουμε το EDF στον προϋπολογισμό. Ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας ε, θα έχει αύξηση 20%. 20,6 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια, τα οποία θα διοχετευτούν στην καταπολέμηση της ε, φτώχειας και σε άλλες δραστηριότητες. Όσον αφορά τη δομή θα βασιστούμε στη τρέχουσα γεωγραφική δομή του DCI. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε στρατηγικούς στόχους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την επιρροή μας στην καταπολέμηση της φτώχειας επικεντρώνοντας την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χρηστή διακυβέρνηση και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα θέλαμε επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στον τρόπο που ξοδεύονται τα χρήματα στα γεωγραφικά προγράμματα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση και να επικεντρωθούμε στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες όπου η επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική μας όσον αφορά τα θεματικά προγράμματα μιλάμε για συγκέντρωση και για απλοποίηση. Θέλουμε να περικόψουμε τα προγράμματα σε μόλις δύο. Το πρώτο θα ε, καλύπτει τα παγκόσμια δημόσια αγαθά, τις προκλήσεις που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βάσει των εσωτερικών της ε, πολιτικών, όπως η κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο καλύπτει ιδιωτικούς παράγοντες. Θέλει να προωθήσει τη δημοκρατία με μεγαλύτερη ένταση, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο δημοκρατικός έλεγχος της εξωτερικής στήριξης θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω πράξεων κατεξουσιοδότηση. Οι πράξεις κατεξουσιοδότηση είναι επίσης απαραίτητες για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει υπογραμμιστεί στη σχετική έκθεση από το Κοινοβούλιο. όπω είπα, η Κομισιόν θα επιθυμεί επίση έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη, Ανάπτυξης. Αξιότιμα μέλη, πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες αυτές χρηματοδοτικές προτάσεις είναι οι σωστές, οι οποίες πλαισιώνουν την ανανεωμένη μας προσέγγιση της συνεργασίας, της αναπτυξιακής συνεργασίας μέχρι το 2020 ενημερώνουν την ε, αναπτυξιακή πολιτική για το μέλλον και αυτό αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια χρυσή ευκαιρία να επεκτείνει το ρόλο της ως παγκόσμιος παράγων και να παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις ε, συνεργατικές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε σχετικά με τα προγράμματά σας. Βεβαίως είμαστε στην αρχή, ε, υπάρχει το Συμβούλιο που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και υπάρχουν και κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το πόσο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ένωση πρέπει να ξοδεύει για την ανάπτυξη στα επόμενα έτη. Έχω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να προβούν σε μία ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και ξεκινώ με τον Φιλίπ Κασπάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίασή του και για όλες τις χρήσιμες ε, πληροφορίες που μας έδωσε διότι όσον αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ε, δίνει μια θετική, δίνει ένα θετικό πνεύμα και διευκολύνει τη συζήτηση. Αντιθέτως όμως την περασμένη εβδομάδα όταν ψηφίσαν την έκθεσή μου και την έκθεση του κυρίου Γκέρενς είχα να αντιμετωπίσω μία στάση λιγότερο αισιόδοξη διότι δύο αυτές εκθέσεις δεν ε, ε, προβλημάτισαν την Επιτροπή μας. Καταφέραμε να επιτύχουμε μια ευρεία πολιτική συνένεση. Ίσως όμως θα έπρεπε να είναι πιο αμφιλεγόμενα και να υπάρχει μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε περαιτέρω διότι ε, ε, περιορίσαμε τη συζήτηση σε μία σύντομη ανταλλαγή απόψεων και πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Δεν ε, με απασχολεί η συνένεση στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Αυτό που με απασχολεί είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου, διότι το γεγονό ότι σήμερα έχουμε περιορίσει αυτή τη συζήτηση σε μία σύντομη παρουσίαση με προβληματίζει γιατί δεν μπορέσαμε όντως να μπορέσουμε να ε, κάνουμε τη συζήτηση όπως θα θέλαμε. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μία καλή συνεργασία και ε, αν θέλουμε να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πρέπει εμείς οι ίδιοι δηλαδή οι βουλευτές να δεσμευτούμε περισσότερο και ίσως ένας τρόπος για να το επιτύχουμε θα είναι να γίνει μια ουσιαστική πλήρη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ναι. Έχουμε ακόμη. Έχουμε περίπου μια ώρα να συζητήσουμε αυτά τα 30 δις συν 24, πόσα, 50, λέει ο κύριος Δίβα. Ναι, καλά τα είπατε. Θα πρέπει να γίνει περισσότερη ανταλλαγή απόψεων ε, και κάποια στιγμή, κύριε Επίτροπε, μετά τις διακοπές. Ίσως θα πρέπει έτσι κανένα δύο ωράκι να τα πούμε όσον αφορά τις δαπάνες αυτών των προγραμμάτων. Να γίνει ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε και ε, τι διαθέσιμα υπάρχουν μετά από τον καυγά με το Συμβούλιο. Δηλαδή, απλώ τις τι πρέπει να γίνει, πέραν να όσων διατίθεται να εκταμιεύσει το Συμβούλιο. Εάν βέβαια θέλετε να έρθετε Και έτσι να έχουμε περισσότερο χρόνο διάθεσή μας για να τα πούμε. Επίτροπος. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ε, γιατί υπάρχει καλό προηγούμενο και αν εσεί θέλετε να με προσκαλέσετε, δεν πάντοτε να ξέρετε ότι έχετε τόση δουλειά και ε, δεν είναι πάντοτε εύκολο να έχουμε ουσιαστική, πολύ ουσιαστική συζήτηση. Πάντως, όποτε θέλετε, όποτε θέλετε να έρθω. Ίσως και ατύπως, γιατί ξέρω ότι το επίσημό σας πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο. Και πολλές φορές δεν μπορείτε καν να υποβάλλετε τις ερωτήσεις που θέλετε και, και, και εμεί έχουμε πολλά να κάνουμε. Αλλά, εν πάση όμω προτίθεμαι να συζητήσουμε όλα τα ενδιαφέροντα που σίγουρα έχετε. Ανά πάσα στιγμή που εγώ βρίσκομαι εδώ. Την περσμένη εβδομάδα, μόλις ήμουν στη Σομάλια, στη Σομαλία, συγγνώμη, στο Τζιμπουδί, δεν ήμουν στη Βρυξέλλας. Να, γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, για τα όσα μας ε, εξήγησα την συντομία για τα σχέδιά σας. Τέσσερα θέματα έχω να θίξω, αν δεν έχετε αντίρρηση. Το πρώτο είναι ότι συζητούμε για χρηματοδότηση, για το μέλλον της ε, ανατησιακής βοήθειας, αλλά πρέπει πάντοτε τα εξή τέσσερα να τηρούμε. Συνέπεια μεταξύ των πολιτικών, ούτω ώστε να μην ε, περιορίζουμε την αποτελεσματικότητά μας, Χρειάζεται συνεργασμό μεταξύ κρατομελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη αποτελεσματικότητα, μην έχουμε επικαλύψει στι δράσει. Επίση, χρειάζεται αποτελεσματική έσπαξη των φόρων από τι αναπτυσσόμενε χώρε και ε, επενδύσει και μεθόδου χρηματοδότηση, το οποίο θα πρέπει να τονιστεί όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συστήματα αποταμίευσης και ασφάλισης τώρα. Στην ανακοίνωση Μπαρόσο, όσον αφορά το πολιετές πλαίσιο του 14 20, μας αναφέρει ότι για να καλύψουμε τις διεθνείς εξελίξεις, η Κομισιόν θέλει να επαναπροσανατολίσει τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σε ε, αναδυόμενες μηχανικά προχωρημένες χώρες και ξέρουμε ότι το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό και θα πρέπει ίσως να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Πώς θα κάνετε αυτόν τον επαναπροσανατολισμό εάν ε, γίνει κατευθείαν κάποια άνοδος χρηματοδότησης προς αυτές τις περισσότερε χώρες, τι θα γίνει τις πέρα από την Κίνα και την Ινδία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ε, έχουμε ευθύνη, δεν μπορούμε να την ε, απεμπολίσουμε. Να γίνει ο επαναφροντισμός των πόρων έτσι, ούτω ώστε οι κυβερνήσει των αδειωμένων κυβερνήσεων να συνειδητοποιήσουν την δική του ευθύνη. Πολύ καλά είναι να μπορεί κανένα να αγοράζει μια τζάγκουαρ σε σχέση με τις χαλιβουργίες μας, αλλά θα πρέπει πριν αρχίσει αυτές τις επενδύσεις ή τις τζάγκορ που αγοράζουν, ας πούμε, να, να κοιτάξουν τι θα κάνουν με, με, αυτού που πεινάνε στη χώρα τους. Κάτι άλλο τώρα. Πριν από λίγο μα αναφέρατε για την ευελιξία. Θέλετε περισσότερη ευελιξία για το πού και πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα. Συμφωνώ και το καταλαβαίνω, αλλά θα ήθελα να μας πείτε κάτι άλλο. Να δεσμευτείτε ξεκάθαρα ότι εκ των προτέρων συμφωνείτε όσον αφορά τους στόχους, αλλά και τις προτεραιότητες που θα προσανατολίσουν αυτή σας την μεγαλύτερη ευελιξία. Τέταρτη παρατήρηση είναι. Ούτε στην ανακοίνωση Μπάραζο, ούτε σε όσα εσείς εισηγηθήκατε, και φυσικά εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν λόγοι για να είσαστε σύντομοι. Δεν είπατε τίποτα για τους πιο περιθωριοποιημένους, τους πιο ευάλωτους σε αυτές τις ε, χώρες. Είτε υποφέρουν από δυσμενείς διακρίσεις, για οποιοδήποτε λόγο. Τέλο πάντων, οι φτωχότεροι των φτωχών σε αυτές τις χώρες. Χρειάζεται η μεγίστερη αποτελεσματικότητα για την δυσιακή βοήθεια ούτω ώστε να μπορέσουν αυτοί να ξεφύγουν από αυτή τη φτώχεια την ε, ακραία που του μαστίζει. Είναι βασικό μα καθήκον. Είναι θέμα δικαιώματο των πολιτών. Είναι θέμα κοινωνική δικαιοσύνη. Μα ακόμα λοιπόν και στις φτωχότατες αυτές χώρε. Κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο για κάποια έργα τα οποία στην αρχή μας φαίνονταν ότι θα συζητούν στο πλαίσιο πράξεων κατεξουδότηση και τελικά δεν καταλήξαμε σε κάτι τέτοιο. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν για τις ε, κατεξουδότηση πράξεις θα ε, κυκλοφορήσει σε λίγο. Είναι σημαντικό να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε επειδή αυτή η συζήτηση αναβάλλεται συνέχεια ε, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω επ' αυτού εάν συμφωνείτε με την αρχή του παραλληλισμού μεταξύ των δύο νομοθετικών οργάνων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποδέχεστε ή μάλλον απορρίπτετε όπως εμείς ε, την ιδέα ότι το Συμβούλιο θα έχει περισσότερο, πιο ισχυρή γνώμη στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο ερώτημα, οι συζητήσεις ε, με την Κομισιόν ακόμη και, ε, και κλεισμένων των θυρών είναι πάντοτε πολύ καλές. Ε, κοιτώντας τον κύριο Δομένικο Χωσό έχω την εντύπωση ότι θέλουν να μας πούνε ότι έχουμε δίκιο αλλά δεν το ομολογούν. Αυτό δεν συμβαίνει. Ε, τότε ίσως δεν κατάλαβα καλά. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τον προϋπολογισμό και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είχαμε μια συζήτηση σήμερα το πρωί, αρκετά ε, λεπτομέρη σχετικά με τη μείωση ορισμένων πιστώσεων από την Κομισιόν. Είπαμε την άποψή μας ε, σε σχέση με αυτή την απόφαση. Θα ήθελα να διευρύνω λίγο το πεδίο σκέψης ε, περί προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ε, αρχικό σφάλμα στις αναπτυξιακές πολιτικές. Όλοι προσπαθούν να επιτύχουν ε, το 0,7% Εάν ε, και οι 27 τηρήσουν τη δεσμευσή τους, τότε οι συμμετοχές θα αυξηθούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναφερόμαστε σε έλλειψη χρημάτων για να αυξήσουμε και να επεκτείνουμε την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Όταν λοιπόν περιοριζόμαστε ε, στα όρια τα δημοσιονομικά της Κομισιόν, οτιδήποτε αφορά το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας υπόκειται στην ίδια αρχή δημοσιονομική όπως και οι διευθύνσει. Πιστεύω λοιπόν ότι ο προπολογισμό πρέπει να αυξηθεί και αυτό θα γίνει όταν θα ενσωματώσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στηρίζω, αλλά θα πρέπει να συγχρονίσουμε την πολιτική βούληση αφενός για εκχώρηση περισσότερων κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και αφετέρου την αύξηση του προϋπολογισμού για την Κομισιόν πώς είναι δυνατόν να έχουμε επαρκή εξουσία επί των 27 άλλων παραγόντων εταίρων μας, εάν εσείς οι ίδιοι μειώσουμε την ε, οικονομική στήριξη σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης ε, το, πρόβλημα, το μελλοντικό πρόβλημα των ΑΚΕ. Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού τις χώρες Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι αμφισβητούμε αυτή τη συνεργασία, αυτή την εταιρική σχέση που κατά την άποψή μου είναι υποδεγματική. Από την άψη της ε, Αφρικής ε, το να υπάρχει αυτή η διασφάλιση ε, κονδυλίων σημαντικών σε πολιετές πλαίσιο και από τη δική μας την πλευρά μας συμφέρει να συνεχίσουμε αυτά τα πλαίσια συνεργασίας ε, πέραν από την αναπτυξιακή πολιτική. Ε, πολλές αφρικανικές χώρες ε, ε, λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Από πολιτική άποψη λοιπόν είναι μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Πιστεύω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη που δεν θέλουν αυτή την πολιτική είναι τα κράτη που δεν θέλουν να αναπτύξουν αυτές τις, ε, αυτά τα πολιτικά πλαίσια βάσει τη Συμφωνίας της Κοτονού. Το τελευταία ερώτηση, η τελευταία ερώτηση ε, ε, σκέφτηκα στο, κατά τη διάρκεια του διαρθρωμένου διαλόγου στη Βουδαπέστη που μίλησαμε για τις τοπικές εξουσίες, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Εξαιρετική ε, συνεννόηση, δεν συμφωνήσαμε στα πάντα, αλλά υπήρξε κάποια ε, σύγκληση. Αυτή, αυτό είναι το τίμημα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα σε αναπτυξιακά θέματα. Ε, νομίζω είχατε ανακοινώσει η παρουσία της κυρίας Κελέρη, η οποία υπήρξε μέλος πολύ ενεργό, ε, μια ανακοίνωση σε σχέση με τον ε, διαρθρωμένο διάλογο και τη συνέχιση αυτής της μορφής διαλόγου. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Επίτροπε, υπήρξαν τρεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Ναι, Όντως ήταν πολύ σοβαρά θέματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω εν το μέτρο του δυνατού. Ουσιαστικά δεν έχω διαφορετικές απόψεις. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή ε, συζητάμε και ε, επεξεργαζόμαστε τις προτάσεις για εφέτος. Ίσως δεν το ανέφερα στην παρουσίασή μου, αλλά υπάρχει μία πρόοδος των εργασιών. Ε, δεν έχω όσον αφορά τις παρατηρήσεις ε, σχόλια, αλλά είναι ένα θέμα πολιτικής. Είδα σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ε, Ιδίω στο Μπαγκλαντές παραδείγματο χάρη, οπότε εξαρτάται και από την κυβέρνηση όσον αφορά τα διάφορα μέσα. Το, μάλλον το εργαλείο ο, συνεργασίας νομίζω ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε χώρα και κάθε χώρα ε, είναι επιλέξιμη για μια τέτοια συνεργασία. Οπότε... Ε, ότι ναι, μεν καταλαβαίνω αυτά τα οποία λέτε για την Ινδία και το, τη Βραζιλία και αυτές οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ε, ε, ανάπτυξή τους για αυτόν τον ε, τον λόγο ε, διότι εμπλεκόμαστε σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως όχι άμεσα αλλά πιστεύω ότι η εμπλοκή μας πρέπει να αποβλέπει ε, στην πρόοδο των χωρών και είναι ένα θέμα φιλοσοφικό διότι όπως σας είπα εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το λαό αυτή είναι η φιλοσοφία μας αλλά για να εφαρμόσουμε τα διάφορα μέτρα απευθυνόμαστε στις χώρες και γι' αυτό πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε να εντοπίσουμε τις πλέον φτωχές χώρες όπου έχουμε περισσότερες δυνατότητες και όπου θα μπορούσε να υπάρξει μία αλληλεπίδραση και επέκταση των επιδράσεων αυτών στις γειτονικές χώρες. Ε, διότι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 191 χώρες εκ των οποίων ίσως 40 ε, είναι αναπτυγμένες, ε, έχουμε ίσως 150 στις οποίες δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και τις 150, πρέπει να καταρτήσουμε μία σειρά προτεραιότητας και γι' αυτό ε, θα ήθελα να σας πω ότι η Κίνα δεν χρειάζεται ίσως αναπτυξιακή βοήθεια σαν χώρα, αλλά τη χρειάζεται σαν λαός. Οπότε αναλόγως των περιπτώσεων θα πρέπει να υπάρξει αναπτυξιακή βοήθεια. Όσον αφορά την περαιτέρω ευαισθησία, θέλω να πω ότι όσον αφορά τις διαδικασίες χρειαζόμαστε διάφορες πράξεις κατ' εξουσιοδότηση και όταν ανακαλύπτουμε κάτι που χρειάζεται να αλλάξει Ίσως είμαστε δεσμευμένοι έναντι της επομένης νομοθετικής πρόπτικης και θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να αλλάζουμε τις καταστάσεις πιο εύκολα. Αυτή είναι η ευελιξία την οποία υπενήσωμε, διότι διαφορετικά πιστεύω ότι θα πρέπει, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άκαμπτο πλαίσιο, δεν πρέπει να ε, είμαι βάλωτος σε οποιοδήποτε πολιτικό λόμπι οι οποίοι θα μου λένε κάνε αυτό ή κάνει εκείνο. Αν μου πείτε <clears throat> φτιάξε δρόμους ευχαρίστως αρκεί να έχω τον προπολογισμό. Αν και είναι μια ε, στενά νοούμενη ε, ενίσχυση αναπτυξιακή στο θέμα αυτό. σχετικά με το τελευταίο θέμα για τα δικαιώματα των πολιτών νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί και γι' αυτό έχω αλλάξει άποψη σχετικά με την βασική στοιχειώδη εκπαίδευση ε, και την βασική υγειονομική περίθαλψη. Δεν μπορεί να υπάρξει ενίσχυση μιας κοινωνίας η οποία δεν έχει πρόσβαση στη ε, βασική εκπαίδευση και στις ουσιαστικές υγειονομικές ανάγκες. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να ε, περιμένει κανείς ότι θα επιτύχει στον τομέα αυτό και έχω πλήρη κατανόηση. Τώρα, σχετικά με αυτό που με ρώτησε ο Τσάρλς, πρέπει να σου πω ότι ουσιαστικά ε, ε υπάρχουν ε, ε, δύο δημοσιονομικές αρχές, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για μένα δεν υπάρχει μία που προηγείται της άλλης. Ε, βεβαίως υπάρχουν και συνθήκες και πρέπει να εφαρμόζω αυτά που λένε οι συνθήκες. Αλλά γενικώς και όσον αφορά το ποια είναι η αρχή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, πρέπει απλώς να ερμηνεύσει κανείς το πνεύμα των λεπτομεριών των συνθηκών και αυτό είναι σαφές γι' αυτό και η πράξη κατεξουσιοδότηση είναι μια τόσο δύσκολη περίπτωση ε, είναι ίσως ε, ένα δώρο παρηγοριάς αλλά ελπίζω ότι θα βρούμε μια λύση και θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις πράξεις κατεξουσιοδότηση ή στους μηχανισμούς και εις, ε, τα συμπεφωνημένα όσον αφορά την χρηματοδότηση. Αντιλαμβάνομαι τι είπε ο Τσάρλς και συμφωνώ και μαζί του, διότι ε, υπάρχει μία συνεχής φύνουσα πορεία και αν δείτε ε, τι, τι προβλέπετε ότι θα γίνει το 2015 και πού θα βρίσκεται το 0,7% ε, θα δείτε ότι θα έχει μειωθεί. Αλλά παρόλα αυτά οι χώρες πρέπει να ε, καλύψουν τις δαπάνες διότι ε, υπάρχουν οι δημοσιονομικές προοπτικές, φορούν να εξοικονομήσουν κάθε δεκάρα αλλά ακόμη και αν μειώνεται το ποσοστό μας, προσπαθούμε αμέσως ε, να το χρησιμοποιήσουμε διότι διαφορετικά μας ε, λέγουν ε, ότι σε μία περίοδο τέτοιας λιτότητος ζητάτε αυξήσεις και πρέπει να μπορούμε να αιτιολογήσουμε κάθε αύξηση και να έχουμε ταπεινόφρονες προτάσεις οι οποίες όμως να είναι συγχρόνως φιλόδοξες. Μπορώ να σας διακόψω. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη πρέπει ε, να κινούνται σωστά και να μας πούνε εάν δεσμεύονται από την ε, υποχρέωση να καταναλώνουν το 0,7% σε αναπτυξιακή βοήθεια το 2015, διότι εδώ είμαστε υποκριτές. Από τη μία πλευρά λέμε ότι το 0,7% είναι η συνένεση και μετά τα κράτη επικαλούνται τις ε, δημοσιονομικές τους δυσκολίες. Ας μας πούν τι γίνεται διότι ορισμένοι ε, σέβονται τους στόχους τους και αναφέραμε σήμερα το πρωί αυτοί, ε, ε, αυτούς οι οποίοι υπερβαίνουν το 0,7 και αυτούς οι οποίοι δεν φτάνουν καν σε αυτό το κατόφλι το οποίο έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Είναι τελείως απαράδεκτα αυτά τα οποία μου λέτε. Εγώ εξακολουθώ να παρακολουθώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπε με τρόπο που με ικανοποιεί ότι η υποσχέση θα τηρηθεί σύμφωνα με το περσινά δεδομένα, δηλαδή το 0,7 είναι εδώ. Και οι χώρες έχουν λάβει δεσμεύση να το επιτύχουν. Δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή πρόοδος, και ορισμένες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν μειώσει προσωρινά. Ε, υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες ε, δεν συμμετέχουν ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτή η λογική του 0,7 είναι σημαντική για την υπερασπισία αυτής της πρότασης. Κατανοώ ότι η ανησυχία σας ε, σε σχέση με τη, ότι η πρόοδος το 2010 σχέση με το 2009 δεν ήταν επαρκής, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπήρξε κάποια πρόοδος, υπήρξε κάποια τάση. Εμείς θα κυκλοφορήσουμε εκθέσεις, θα πιέσουμε και θα συνεργαστούμε με τις χώρες. Δεν είναι χαμένη υπόθεση θα έλεγα. Καταλαβαίνω τη φιλοδοξία, ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά το κοτονού. Κατά την άποψή μας ε, βρισκόμαστε σε περίοδο προβληματισμού επειδή το 2020 είναι το έτος λήξης. Θα πρέπει να προβληματιστούμε. Εξακολουθεί να μην μου αρέσει η συζήτηση που είχαμε με τον Μάικλ για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Προσπάθησα ό,τι μπορούσα και ήμασταν εξαιρετικά ευέλικτες στις προτάσεις μας. Προσπαθούσαμε να μειώσουμε κάποιες φιλοδοξίες ε, καταλαβαίνοντας τις δυσκολίες αλλά δεν λειτουργήσε επειδή μερικές ε, χώρες υπήρξε κάποια παρανόηση και είναι σημαντικό και η άλλη ομάδα, οι εταίροι μας να προβληματιστούν ε, σχετικά με αυτή την εταιρική σχέση. Δεν είναι δυνατόν ο μικρότερος παρονομαστής ε, τη σχέση μας με την ομάδα και να καθορίζει τη σχέση μας με την ομάδα και Σήμερα απογοητεύτηκα με, για τις διαπραγματευτικές μου ικανότητες, επειδή δεν καταφέραμε να επιτύχουμε έστω και κάποια μικρή εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αλλά η πρόταση ήταν πολύ ελαφριά όχι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Πιστεύω ότι απορρίφθηκε με τρόπο άδικο. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε έκκληση στους εταίρους μας να ε, σκεφτούν αυτή τη, να προβληματιστούν για αυτή την εταιρική σχέση. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και έχουμε μία περίοδο 7 ετών, μεγαλύτερη μάλιστα, να δούμε πώς θα προχωρήσει ο πολιτικός διάλογος με τους συνεργάτες μας. Εάν αυτοί δεν έχουν τη διάψη θα πρέπει να το εξετάσουμε. Υπάρχουν οι δομέ για να το κάνουμε αυτό. Είναι μια καλή λοιπόν περίοδος για προβληματισμό και από τις δύο πλευρές. Και τέλος, σε σχέση με το διαρθρωμένο διάλογο, πιστεύω ότι ήταν επιτυχής. Πολλά στοιχεία θα συμπεριληφθούν στην πρόταση μηχανισμού και η ανακοίνωση θα κυκλοφορήσει του χρόνου. Θα συμπεριληφθεί λοιπόν, δεν υπάρχει καμία διαφωνία εδώ στο δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους. Um, using my privilege as chairman, I just want to... πρόεδρος θα ήθελα να επισημάνω ότι καθώς εμείς ε, συζητάμε για αυτές τις τεράστιες ποσότητες χρημάτων, μόλις ακούσαμε ότι η Ιταλία αυτή τη στιγμή ε, δέχεται επίθεση από δημοσιονομική άποψη και η Ισπανία από όσο φαίνεται επίσης καθόμαστε και μιλάμε για αύξηση της αναπτυξιακής αρρωγής προς τους στοχότερους από 17 δισεκατομμύρια σε 20 δισεκατομμύρια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Στήριξης και, από 20... και σε 22 εκατομμύρια στο πλαίσιο του EDF. Θα πρέπει να μπορέσουμε αυτό να το πουλήσουμε σωστά, να το διαφημίσουμε σωστά στους ε, σε όσους μας έχουν εκλέξει. Ε, έχουμε την ελληνική κρίση, την ιταλική, την ισπανική ίσως. Ε, δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι πώς θα πείσουμε για αυτές τις τεράστιες χρηματικές ποσότητες στο το εκλογικό σέμου. Ε, παρακαλώ. Οι συντηρητικοί στη Βρετανία θέλουν να χτυπήσουν, ε, το, να ισχύει την εξουσία του ε, των χρηματαγορών. Θα ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω την κυρία Κέλλερ και μετά τον κύριο Πάλμερ. Αλλά πρώτα απ' όλα, θέλετε να απαντήσετε ήθελα να πω προς το Ηνωμένο Βασίλειο ότι το κοινοβούλιο σας ε, ζήτησε να αυξάσετε ε, την αναπτυξιακή βοήθεια. Λοιπόν, ίσως πρέπει να πείσετε τη Γερμανία, η οποία δεν αντιμετωπίζει δημοσιονομικές δυσκολίες και δεν κάνει τίποτα να αυξήσει το προϋπολογισμό της. Ναι, το ο κόμμα μου αύξησε τη βοήθεια με τα μεγάλες δυσκολίες για να πει στους άλλους. Θα ήθελα όμως εδώ να σας πω κάτι ότι το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όντως ε, είπε ορισμένα πράγματα αλλά όσον αφορά τα δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια για τα οποία συζητάμε όντως ε, έχουμε, κάνει, έχουμε διαθέσει 40 δισεκατομμύρια ε, τα οποία δώσαμε σε ένα κράτος μέλος και ενδεχομένως θα δώσουμε και σε άλλο. Βοηθάμε ε, χώρες εντός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσά τα οποία ε, ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα οποία θα χρειάζεται ο υποανάπτυξη κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο Λόρδος Ντόμπς ο οποίος είναι εδώ και είναι ε, ένας γνωστός συγγραφέας ε, ο οποίος ε, μας παρακολουθεί. Ναι, η Φραντσέσκα. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να αναλάβω τις ευθύνε μου για τη χώρα μου, τη Γερμανία, αλλά πρέπει να δούμε ότι αν δούμε από πού βρίσκουμε τα χρήματα, θα δούμε και από πού προέρχεται η η ε, φορολογία και έχουμε έναν υπουργό ο θέλει να φύγει από το Υπουργείο μας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και πρέπει να σας πω ότι επιπλέον έχουμε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των κλιματολογικών αλλαγών οι οποίες λέγεται ότι είναι διαφορετικές και θα έπρεπε να αλλάξουν και ενδεχομένως θα πρέπει να τεθούν ορισμένα κριτήρια. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ε, επιβεβαιώσουμε και να δούμε ότι πρόκειται για μια χρηματοδότηση η οποία συμπληρώνει τα ε, ισχύοντα μέτρα χρηματοδότησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση ε, δεν ε, συνδέεται άμεσα με ε, τον προϋπολογισμό αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε για οποιοδήποτε είδος το οποίο υπάρχει γιατί ορισμένοι ε, χρησιμοποιούν το περίπλοκο σύστημα με τη δεσμευμένη βοήθεια και τη μη δεσμευμένη βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η νέα αναπτυξιακή πολιτική που πρεσβεύεται και πώς ε, σκοπεύετε να προβείτε σε διαβουλεύσεις για την ε, νέα στρατηγική. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε Ξέρω βέβαια ότι η Ντεύκο έχει ε, πολύ δύσκολο έργο εδώ, αλλά πρέπει να δούμε ε, τι, πού μπορούμε να παρέμβουμε και ποια είναι τα άλλα θέματα διότι σε πολλά θέματα δεν προχωρούμε ε, σωστά και πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να ε, προχωρήσουμε διότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στις ανησυχίες μας. Πώς μπορείτε να παρέμβετε λοιπόν για να επιτύχετε αυτή, αυτό το σεβασμό. Επίσης αναφερθήκατε ε, στα χρήματα που αποδίδουν, value for money. Οπότε ε, ζητάμε να αποδίδουν περισσότερο τα χρήματά μας. Αυτό θέλει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα σχολεία ασχέτως του επίπεδου της παιδείας και στη Γερμανία παραδείγματος χάρη προσπαθούμε ε, να δημιουργήσουμε μία κατάσταση όπου πρέπει να δούμε ε, πώς ε, εσείς τοποθετήστε στις νέες συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται και εν ώψη του Πουσάν όπου πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά θα επανακύψουν δηλαδή όταν μιλούμε για value for money για απόδοση των επενδύσεων δεν αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση του Παρισιού αλλά σε μία τελείως διαφορετική κατάσταση. Και ε, θα ήθελα τώρα όσον αφορά το νέο μέσο για την Αφρική να μου πείτε πώς αυτό συνδυάζεται με τα άλλα ισχύοντα προγράμματα. Τι μορφή θα έχει και ενδεχομένως μπορείτε να μας πείτε αν ε, ε, είπατε ότι η αναπτυξιακή ευρωπαϊκή πολιτική και το σχετικό ταμείο θα ε, παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως μπορείτε να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει όλο το σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Επίτροπο για την παρουσίαση του και τις επεξηγήσεις που έδωσε. Χαίρομαι που στην ανακοίνωσή της ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Κομισιόν δηλώνει ότι υπάρχει δέσμευση για 0,7% στην αναπτυξιακή συνεργασία και ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Ωστόσο, κύριε Επίτροπε, Θεωρώ ότι είναι δυστυχές ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι οι συνθήκες ε, δεν πληρούνται για την υλοποίηση. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι αυτό θα επέτρεπε αυξημένο δημοκρατικό έλεγχο και αυτό θα επέτρεπε οι συμπολίτε μα να υποστηρίξουν την πολιτική και τι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αναπτυξιακά. Όσον αφορά τους πόρους ε, μιλάμε για 321 εκατομμύρια όπως γνωρίζετε αυτές οι χώρες δεν προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φτώχεια αλλά να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την περιφερειακή τους ένταξη είμαι βέβαιος ότι ένα αντόκ ε, ε, χρηματοοικονομικό σύστημα για σπίτι ΟΕΜ θα τους επιτρέψει να υπάρξει μια πραγματική εταιρική σχέση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε, στην, να βασιστούμε στην υποστήριξή σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν αντιπαθεί την αναπτυξιακή πολιτική, αλλά οι τράπεζες ε, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πούμε στους πολίτες αν θα επιλέξουν να δώσουν τα χρήματά τους για να βοηθήσουν τη φτώχεια στο τον κόσμο. Η συζήτηση αυτή θα αποτύχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την παρουσίασή του και να, να τον συγχαρώ για, την ε, για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Και έτσι ελήφθησαν όλες αυτές οι προτάσεις για την αύξηση ε, του κεφαλού 4 των πόρων, για αυτές τις δράσεις της Ένωσης, όλα τα θέματα του να καλυφθεί ευελιξία, Επίσης, για παράδειγμα, αυτό το δικό αποθεματικό για, το, την κρίση στο γεωργικό τομέα, για αυτά τα 500 εκατομμύρια ή και επίσης εκεί που ρητός προβλέπεται ο ενδεδελχέστος έλεγχος του Κοινοβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Επομένως, αυτά έχω να σας τα πω ότι με απασχολούν και μου αρέσει πάρα πολύ ο αυτή η θέσπιση του φόρου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών για το 2018. Επομένως, μια σύντομη σκέψη με τον αυτή. Θα ήθελα να πείτε κύριε Επίτροπη για τις ε, προκλήσεις που έχουμε. Έχουμε αυτό το 0,7% και σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας και πρόκειται για τον συντελεστή που είπαμε ότι προβλέπεται για το 2015, κάτι το οποίο συνδέεται με τους νέους στόχους Οπότε είναι ε, ένα κάβος που να τον περάσουμε, ε, στόχος για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει μετά το 2015 να αρχίσουμε από τώρα να σκεφτόμαστε τι γίνεται σε σχέση πάντα με τους στόχους της χιλιετίας που ήδη έχουμε προγραμματίσει. Οπότε αυτό έχει σχέση άμεση με την εκρίζωση της φτώχειας και την καταπολέμηση του κλίματος, της αλλαγής του κλίματος και ξέρετε Επίτροπε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και ε, εάν θέλουμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε κάποιες ε, ζώνες ε, στον κόσμο συντονισμένο. Οπότε αυτό το οποίο με απασχολεί και το οποίο άμεσα συνδέεται με την πρώτη σκέψη την οποία σας ανέφερα είναι το εξή. ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις αναδυόμενες χώρες και θα πρέπει πώς ταυτόχρονος να δούμε τι θα γίνει με τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν είναι δυνατόν την ύφη για την κρίση να την πληρώσει η πολιτική της συνεργασίας με κάποιες χώρες στρατηγικής σημασίας για τη σημερινή συγκυρία για τη συνεργασία των μερών για κάποιες χώρες οι οποίες ακριβώς τώρα έχουν αρχίσει να, να, να, να εισφέρουν ε, χρήμα, να βοηθούν ε, όλο τον κόσμο και εμείς δεν μπορεί να τις εγκαταλείψουμε σε, κάπου, σε μια τόσο σύντομη, ε, συγγνώμη, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Ευχαριστούμε λέει ο κ. Λίβα και δίνει τον λόγο στον Επίτροπο. Πίμπαλξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσω με τα όσα ανέφερε ο κύριος Κάσμαν για την αναλογία που πάει εις στους καταναλωτές στην ανάπτυξη γιατί θα πρέπει κανείς να διδάξει μεγέθους τι έγινε για μια τα αιτία και τι καταφέραμε τόσο σύντομα. Όχι, όχι, δεν, δεν έχουμε εδώ πέρα υπερακοντήσει στο στόχο διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι θέλει ο κόσμος, να δει ε, η οικογένεια, η δομή της κοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντικά, άνοιγμα στον κόσμο και άρα να βοηθάμε ουσιαστικά όταν χτυπάει η τραγωδία. ρύζι, καλαμπόκι. Αυτό δεν είναι μόνο, δεν, είναι, δεν κανεί σε αυτό. Και το είπε και στη διάσκεψη ο Κάμερον. Εδώ και τώρα θα πρέπει να δοθεί βοήθεια και κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να έχουμε μια σωστή αναλογία στις προσπαθίες μας. Νομίζω ότι ακόμα απομένουν πολλά να κάνουμε για τους φτωχούς, τους φτωχότερους στον κόσμο. Επομένω, δικαίω αυτοί έχουν κάποια πικρία εστραμμένη προς εμά Αυτά όσον τι τις και κάποια στιγμή θα δούμε τι θα κάνουμε και για τη Σομαλία όπως και κάναμε, όπως και στο, στο Αφγανιστάν που πολύ περισσότερα δώσαμε. Δώσαμε περισσότερα από όσα αν ήμασταν σε αναπτυξιακή δράση. Αυτό δεν πάει να πει ότι κάνουμε λάθος. Αλλά έτσι είναι. Και εχουν δυο δύο-τρει προκλήσει σε παγκόσμια κλίμακα. Ασφάλεια, διατροφική. Και για την κλιματική αλλαγή. Στη Σομαλία, στο Τζιμπουτί. Ε, δεν έχουν αφάνα, δεν έχουν νερό. πώς θα τους βοηθήσουμε και αυτό που θα γίνει μόνο μια σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης, την οποία και θα βοηθήσουμε. Επομένω, θα είναι πάρα πολύ απόδεινο το να φύγουμε το 0,7. Δεν από τα κονδυλία μας στους 27. Κοιτάμε τις πληρωμές, τον προπολογισμό και η Λετωνία και η Μάλτα δίνει την εισφορά της. Η Πολωνία συμμετέχει. Να, η διαφορά. Είναι μια κοινή δραστηριότητα, δεν είναι, δεν είναι συγκερασμός ατομικών δραστηριοτήτων. Όλοι μετέχουν. Άρα, έτσι θα εξασφαλίσουμε κάποια αποτελέσματα. Στου Μαγκλαντέ, εμφύλοι πόλεμοι, Πακιστάν, δύσκολε περιπτώσει. Καλά, καλά, θα πρέπει και προσπάθεια να διέπεται από αναλογία. Τι να κάνουμε για το Πακιστάν, να το αφήσουμε όσο έχει. Μα τότε θα έχουμε ανθρωπιστική τραγωδία. Άρα, στρατευόμαστε και στηρίζουμε. Συζητάμε την πολιτική, ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, περιορισμό υγείας, παιδείας κλπ. Άρα όλα αυτά στέκουν. Για την προσθετικότητα, από ό,τι ξέρω, η Επιτροπή δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ένα μέρος της αντιστοιχικής προσπάθειας όντως θα πρέπει να επικεντρώνεται στην μείωση του κινδύνου, στην αλλαγή του κλίματος. Καρεβική και ειρηνικό εννοώ. Τα σχετικά κράτη εκείνα ποτέ δεν θα έχουν αρκετή ικανότητα να προστατευτούν κατά των θεομηνιών, κατά της αλλαγής του κλίματος. Υπάρχουν οριζόντιες δραστηριότητες βέβαια. Ο ΣΑ κάτι κάνει από ό,τι μου λένε και ότι σύμφωνα με τις στατιστικές και επίσης δεν είναι πολλά τα λεφτά, 50 εκατομμύρια μιλάμε για την περίοδο 10-12. Τι θα γίνει τώρα, τι να σας πω. Ελπίζω να κάνει το G20 ό,τι έχει πρεσβεύσει η Γαλλία, το Βέλγιο έχει δεσμευτεί και άλλοι συνάδελφοι μου λένε ότι θα υπάρξει κάποια χρηματοδότηση σταθερή όπως χρειάζεται. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει πίεση να βγουν από εκεί κονδύλια να πάνε κάπου άλλο. Δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν, δεν, δεν υπάρχει λόγος το 07 να σπάσει τα δύο. Τώρα για την ε, βοήθεια. Δεν είναι ψευδής πόδι. Πόθη. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Η συνθήκη έχει θέσει την εκρίζωση της φτώχειας σαν ε, στόχο. Έχουν τεθεί στόχοι, μελετώνται οι προσπάθειες, τα αποτελέσματα. συνεργασία με την εκαστοτε χώρα, στήριξη από την κυβέρνηση και ανάληψη δράσης ή αντίδρασης σε περίπτωση προβλήματος των ανθρώπινων δικαιώματων όπως γίνει Γιατί θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορούμε να λάβουμε δράση οι εταίροι μας. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη σχέση, πολιτική σχέση, Πότε δεν έχω πει ότι θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στις περιπτώσεις που κάποια κυβέρνηση βάζει κόσμο στη φυλακή. Οπότε δεν ούτε, ούτε καν λέμε αν το κάνετε αυτό θα πάρετε τα χρήματα. Συνήθως έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για τη συγκεκριμένη χώρα. Δεν νομίζω ότι δεν τρέχουμε κίνδυνο να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Όχι, όχι, δεν έλεγα για τέτοιου είδους ε, προϋποθέσεις στην ε, ανάπτυξη. Εγώ έλεγα το ότι δίνουμε χρήματα για να φτιάξουν δρόμο, όμως, τα θα πει ότι δίνει κανεί τα χρήματα, αλλά λέει θα χρησιμοποιήσω όμω για το να φτιάξω τον αυτοκινητόδρομο εταιρεία τη δική μου χώρα. Όχι, όχι, όχι, λέει ο Επιτρόπο. Από ό,τι ξέρω ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν έχουν γίνει τέτοια πράγματα ή στι χώρε τη Ένωση. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία για διαζωογονισμούς. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Δεν πάνε στην Αιθιοπία οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Προσπαθούν να τις φέρουν, αλλά δεν πάνε. Έχουν τόσε καλές δουλειές στην Ευρώπη. Επομένω. το αποτέλεσμα τι είναι, πάνε Ινδοί, πάνε Κινέζοι και κερδίζουν διαγωνισμό. Καταλαβαίνετε. Σε σχέση με αυτό, ποτέ δεν έχουμε πει. Θα πάρετε τα χρήματα μόνο αν κάνετε κατέ. Πότε, από ό,τι ξέρω, πότε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα τον κοιόμαι. Βάλει φορμάνι τώρα, να πιάσουν το, τα χρήματα μα. Είναι σχήμα λόγου. Και έχει σχέση με το πρώτο μα θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να φτιαχτούν σχολεία ανεξαρτήτω του αν υπάρχουν μαθητές. Όταν φτιάχνετε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το τι προκοδότηση υπάρχει, τι θέλει κανείς να πετύχει. Ακούγεται σκληρό, αλλά ε, δεν είναι αυτό που φαίνεται το να πιάσουν τόπο τα χρήματα, στο value for money προσπαθούμε να πετύχουμε κάποιο είδου ε, μεταβολή προς το καλύτερο, ποσοτική, ποιοτική και ε, έτσι είμαστε πιο στοχοθετημένοι κατά κάποιο τρόπο, πιο εστιασμένοι την προσπάθειά μας. και τα κάθε φορά κριτήρια θα πρέπει να είναι εύστοχα, εντάξει. Αυτό, αυτό προσφέρουν όλε οι χώρε μέλη. Και έτσι, να μην υπόψη ότι ποια χώρα με το οποίο συνεργαζόμαστε, τι προβλέπετε διεθνώ. Για την Αφρική. Για την Αφρική. Έχουμε αυτή την πρόκληση. Μια αυταετία. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, πολιτική γειτονίαση, διάφορα. Με διάφορα πράγματα του έχουμε πλαισιώσει και θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει η ολοκλήρωση και οι δυνάμει που θέλουν την ολοκλήρωση γιατί την υποστηρίζουμε, γίνει πιο ισχυρή και το με, τα, με τις συμφωνίες της DCI, αυτό το να κάνουμε. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις πανεφρικανικές προσπάθειες. Τόσο ό,τι δεν καλύπτεται από το Ταμείο Ανάπτυξη. Είναι κάπως ε, άδικο βέβαια να μην εγκαλύψουμε και την Βόρεια Αφρική. Γιατί για μένα είναι Αφρική και η Βόρεια Αφρική. επομένως θα πρέπει να το λαμβάνω υπόψη, είναι ένα μόνο στοιχείο σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες ιδιαίτερες σχέσεις με την Αφρική, στρατηγικές. Τώρα έχουμε και άλλες ερωτήσεις που άκουσα. Δεν ξέρω τώρα αν σας απορρίτευσα, αλλά για να σας παρηγορήσω έχω να σας πω ότι 27. Τα έχουμε συζητήσει. Υπάρχει κονδύλι για τις χώρες αυτές που θέλετε. Τελικά, υπάρχουν τα μέσα πολιτικής και υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Προτάσεις δεχόμαστε επικοδομητικές, είμαστε ανοιχτοί. Θέλουμε επομένω να κάνουμε κάτι για τις υπερπόντιες χώρες και δάφη. Τώρα, για την ένταξη στον προπολογισμό αυτών των πόρων των αναπτυξιακών του Ταμείου, Είναι κάτι βέβαια το οποίο έχει σχέση και με τους εταίρους μας στην Κοτονού. Υπάρχει ο μηχανισμός αναθεώρησης, είναι πολυμερή συμφωνίες. Και επομένως όταν έχουμε βρει ένα μηχανισμό που αποδίδει, γιατί να τον διαλύσουμε. Μιλάμε για 77 εταίρους. Ναι κύριε Κέλλερ. Αυτό που είπατε ισχύει. Και προσπαθούμε όλα αυτά στις συμφωνίες DCI να τις ε, λάβουμε υπόψη. Τώρα, ο κύριος Κορτές. Τι θα γίνει μετά το 2015. Γιατί Νομίζω ότι αυτή η πολιτική ε, για τη χιλιετία είναι η κινητήρια δύναμη σε όλες μας Νομίζω είναι σωστοί οι δείκτες, τα κριτήρια που έχουμε. Θα συνεχίσουμε τη ρότα αυτή και θα είμαστε και όσο γίνεται ε, φιλόδοξοι. Όχι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα. Δεν είναι δυσνόητο. Είναι εύχριστο. Απλό. Ίσως δεν είναι τέλειο. Για την αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη βιβλική κοινότητα. Θα προσπαθήσουμε να ληφθεί υπόψη ε, η πολιτική για το κλίμα σε όλες τις πολιτικές, διατροφική ασφάλεια, προσφορά ενέργειας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κλίματος. Άρα, με συγκεκριμένους τρόπους, βοηθώντας τις αντισόμενες χώρες. Συνεργασία με τις αντιστοιχομένες χώρες, με πρόκληση. με την Κίνα, ας πούμε. Προβλέπεται αμοιβαία βοήθεια. Η Κίνα είναι από χώρα. Ταυτόχρονα όμως είναι διαφορετική περίπτωση λόγω της, του Άρα, ναι, να λάβουμε τέτοιες δραστηριότητε, αλλά κυρίω θέλουμε να πλησιάσουν περισσότερο τις ΥΠΑ που είναι σημαντικός εταίρος και Υπάρχει γλώσσα επικοινωνία όσον αφορά την πολιτική τώρα, ιδίω επί κυβέρνηση Δεν έχουμε ιδεολογικέ διαφορέ. Επομένω, έτσι θέλουμε να συνεργαστούμε. Έχουμε χαρτιπορία επίση για πέντε χώρε για την ε, βοήθεια, την ε, βοήθεια και επίση έχουμε και μια κοινή πλατφόρμα για παγκόσμια θέματα υγεία. Κατάλαβα που το πάτε. Νομίζετε ότι έχουμε γίνει ουρά. Τον είπα. Εμείς όμως θεωρούμε ότι 80% είναι η ανάπτυξη που βοηθούμε όλοι. Επιτόπου για και στην Αφρική και στη Γάζα. άλλα υπέρ έχει ο καθένα, αλλά κατά επομένω ο ένα συμπληρώνει τον άλλο όσο με αυτό τη είπα. Επομένω. Κίνα, Βραζιλία, που θα δούμε και εκεί, Ινδία, άλλο μέτωπο. Αλλά είναι δύσκολα. Γιατί θεωρούν ότι ανήκουν σε άλλη διαφορετική κατηγορία. Επομένω, ε, η συνεννόηση δεν είναι όσο καλή θα μπορούσε να είναι. Είναι εφιάλτης. Έχω τέσσερις ομιλητές και πρέπει να κάνουμε και τις ερωτήσεις εντό πέντε λεπτών και να απαντήσει ο Επίτροπος. Ε, συγγνώμη, αλλά θα περιορίσω το χρόνο των ερωτήσεων αναγκαστικά σε ένα λεπτό ανά άτομο. Γκάμπι, ο κ. Κάσμαν, Φιώνα και Μικελάντζελο. Δεν θέλετε, όχι, ωραία. Τρεις ομιλητές, λοιπόν, ένα λεπτό ο καθένας, τρία λεπτά συνολικά. θα, θα αποφύγω ορισμένε ερωτήσει γιατί κάποιε έγιναν ήδη. Θα ήθελα συνεπώ να αναφέρω ένα. Να, ζητήσω κάποιε λεπτομέρειε για ένα σημείο. Εγώ δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι αφενό λέμε ότι απέχουμε πολύ από το ε, ε, ε, πρώτο ε, στόχο της χιλίτιας το 2015. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, η καγκελάριος ε, επισκέφθηκε χώρε αναπτυσσόμενες στην Αφρική. Χρειαζόμαστε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική. Η κλασική πολιτική έχει ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο. Τα οικονομικά συμφέροντα τίθεται στο παιχνίδι. Πρέπει να ανταγωνιστούμε την Κίνα δεν είμαστε σε... πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το AIDS. Ήθελα να ξέρω έτσι λοιπόν ποια είναι η θέση των κρατών μελών και αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο στο Συμβούλιο, αν υπάρχει κάποιο κοινό πρόγραμμα για το μέλλον ε, στο οποίο θα επικεντρωθεί η αναπτυξιακή πολιτική. Διαπιστώνουμε ότι για πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις. Κάνουμε έκκληση δηλαδή σε τρίτους, ειδικά όσον αφορά τα επιστημιστικά προγράμματα. Ήθελα να μάθω ποιος είναι ο ρόλος όπου μέσα στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, ε, που διαδραματίζουν στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ορισμένα έργα φροντίζετε, παρακολουθείτε ε, αυτό που γίνεται, παρακολουθείτε εάν υπάρχει αρκετή διαφάνεια ώστε και σε αυτή την περίπτωση να μπορούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις και όχι να ε, δέχεται να τις επιβάλλουν ε, τα οικονομικά συμφέροντα. Μιλήσατε για δύο λεπτά τώρα. Είναι αδύνατο, είναι παράδεκτο να καθόμαστε εδώ ως μέλη ενώ αναλώνεται ο χρόνος από άλλους χωρίς να σας ενδιαφέρει καθόλου ε, τι κάνουν τα μέλη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα και δεν μπορώ να το συζητήσω σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε λίγο χρόνο και η Κομισιόν θα επανέλθει. Ε, θα το συζητήσω με την ε, Κομισιόν. Φιώνα. Τρία γρήγορα θέματα. Πρώτα απ' όλα η νέα ε, κυβέρνηση ε, προστατεύει ε, τον ε, προϋπολογισμό τον αναπτυξιακό από περικοπές όσον αφορά τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ελέγχους ε, με εγγράφων μεμονωμένων χωρών, εγγράφων στρατηγικής μεμονωμένων χωρών. Επίσης, στο παρελθόν μιλήσατε για τη σπουδαιότητα της πρόσβασης στο ηλεκτρικό ρεύμα για όλους. Ε, σαφώς ε, αυτό κοστίζει πολύ και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί χρηματοδότησης για να επιτευχθεί. Αναρωτιέμαι αν έχετε προβληματιστεί περαιτέρω για το ποιοι μηχανισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάτι τέτοιο και για το αν υπάρχουν τρόποι χρήσης του ε, αναπτυξιακού προπολογισμού ως καταλήτη για να ε, υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ναι, ευχαριστώ. Ε, για την πρώτη ερώτηση όσον αφορά το 07 του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Πιστεύω ότι η κατάσταση φέτος θα είναι πιο δύσκολη. Οι βασικές σχέσεις και η στάση του κόσμου και των κυβερνήσεων ως προς την αναπτυξιακή αρρωγή είναι μάλλον θετική. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν όλοι το θάρρος να το πάρουν σοβαρά και αναβάλουν τις αποφάσεις. Αυτό ε, δυσκολεύει τα πράγματα. Αλλά σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τώρα που υπάρχουν τα, συμβουλία του, το συμπεράσματα του Συμβουλίου, ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ε, θα ήθελα να έχουμε επιτύχει όλους τους ε, στόχους της χιλιετίας έως το 2015. Φυσικά αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να μην τα παρατήσουμε όσον αφορά αυτούς τους στόχους για τις ιδιωτικές ε, και δημόσιες ε, εταιρικές σχέσεις. Δεν το στηρίζουμε ιδιαίτερα στην Κομισιόν, το προσπαθούμε επειδή υπάρχει το πρόβλημα της, του υπόλογου, ότι κάποιοι είναι υπόλογοι για τα ποσά το ελεκτικό συνέδριο θα ψάχνει, θα ερευνά πάρα πολύ για τον τελικό αποδέκτη. Προσπαθούμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα για το η πράσινη οδό στην Τανζανία. Κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά στο παρόν στάδιο δεν έχουμε βρει ακόμη μια καλή απάντηση λόγω της ε, ε, ευθύνη που υπάρχει όσον αφορά αυτά τα κονδύλια. το να έχουμε ευκολίες επενδυτικής, επενδυτικές στη Βόρεια Αφρική για παράδειγμα αυτό ξεκινάει και λειτουργεί καλά είναι ένα καλό έργο για παράδειγμα ε, για την αναπτυξή της αιωλικής ενέργειας αλλά δεν είναι ακριβώς συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι λίγο διαφορετικό Όσον αφορά τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το σχεδιάζουμε επειδή τα έγραφα στρατηγικής των χωρών ε, θα πρέπει να είναι μια θεσμικά σωστή πρόταση. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Εγώ είμαι απλά ένα μικρό κομμάτι όλων αυτών των ε, σχέσεων μεταξύ των οργάνων. Ε, δεν φοβάμαι κανέναν έλεγχο τον οποίο κανένας και ειδικότερα οι δημοσιονομικές αρχές θα ενδεχομένως αποφασίσουν. Θα πρέπει να συμφωνηθεί ο χρόνος φυσικά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Σε επίπεδο θεσμών είναι πολύ πιο περίπλοκο όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο και το Συνοβούλιο και οι σχέσεις τους. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ελέγχου και τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, Προσπαθούμε για αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό κοστίζει πάρα πολύ. Οι Αμερικανοί φίλοι μας έχουν τη φιλοδοξία να φτιάξουν ένα δίκτυο στο Αφγανιστάν το οποίο θα κοστίσει τρομακτικά πολύ, είναι πολύ φιλόδοξο το σχέδιο επικροτώ το θάρρο του, αλλά είναι εξαιρετικά ακριβό. Εμεί δεν προσπαθούμε για κάτι τόσο ακριβό. Πιστεύω ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει με έργα μικρότερη κλίμακα και ξέρω ότι κράτη-μέλη όπω η Γερμανία συμμετέχουν σε αυτό για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια βάσει ηλιακών κυψελών. Δεν υπάρχει τεράστια ζήτηση η ζήτηση σε αυτά τα μέρη δεν είναι τεράστια. Έτσι τα κόστη είναι μικρότερα από αυτά που πιστεύει ο κόσμος. Επίσης η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποκεντρωμένο τρόπο θα βοηθήσει κάθε νοικοκυριό να έχει, πρόταση, να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν ξέρω πώς θα είναι δυνατόν να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν θα είναι πλέον απαραίτητο. Μπορεί κανείς να το κάνει φτηνότερα. Ευχαριστώ Επίτροπε για το χρόνο που περάσετε μαζί μας και μην φοβηθείτε να ξανα, μας ξαναεπισκεφθείτε για περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε και άλλα ε, σημαντικά ζητήματα και τις λεπτομέρειες που θέλουμε να συζητήσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε αυτή την επιλογή. Είμαι βέβαιος ότι ο Μάικλ Κάσμαν θα συζητήσει κάποιους από τους ενδιασμούς του ξέρω ότι το πολεμάει και τον υποστηρίζω 100% διότι εδώ δίνουμε χρήματα σε ανθρώπους που χειρίζονται διάφορους ανθρώπους με διακριτικό τρόπο και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και που ανταλέξετε απόψεις μαζί μας. Everybody's Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, τώρα που θα παραμείνουν μόνο όσοι είναι απαραίτητοι σε αυτή την αίθουσα που έχουν παραμείνει, επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Το σημείο 9 της ημερήσιας ε, διάταξης και έχω την τιμή να προεδρεύσω γιατί δεν υπάρχει κανένας πρόεδρος σήμερα αυτή τη στιγμή. αλληλευτικέ δυνατότητε και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται για τη Συμφωνία αλληλευτική Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Κροτηρίου. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης που έχει με εξαιρετική η ικανότητα ε, συνταχθεί από τον συναδελφό μας, τον κύριο Τσάρλς Κέρενς, ο οποίος θα λάβει και το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ που με παρουσιάζετε ε, τόσο όμορφα θα σας πω ότι έχω κάποια κενά όσον αφορά τις ε, γνώσεις για την αλληλεία, ωστόσο είχα την ευκαιρία να συζητήσω με το Πράσινο Ακροτήρι, μια χώρα που διαθέτει πόρους ε, πολύ σημαντικούς ε, και ένα από τα μεγάλα προβλήματα αυτής της χώρας είναι ότι δεν καταφέρνει ακόμη να παράγει την απαιτούμενη ποιότητα προϊόντων ώστε να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το ζήτημα είναι δηλαδή να επιτυγχάνεται η προσταμινεξία στην ίδια τη χώρα. Αυτές οι ληφτικές συμφωνίες έχουν ένα χρηματικό αντίτιμο το οποίο είναι επικερδές για τις ε, ε, χώρες που το λαμβάνουν. Ωστόσο θα κέρδιζαν περισσότερα αν βελτίωναν τις μεταπητικές τους διαδικασίες και αν μπορούσαν να τηρούν το σύστημα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωτόκολλο της Αλληλευτικής Συμφωνίας Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακροτηρίου θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2011 και το νέο πρωτόκολλο θα καλύψει μια τρίτη περίοδο. Η εξουσία μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ε, μπορούμε είτε να το εγκρίνουμε είτε να το απορρίψουμε. Σύμφωνα με το σχέδιο γνωμοδότησης για το οποίο είμαι εισηγητής, ε, χρειάζεται να καθορίσουμε ένα πλαίσιο συνεργασία που θα διευκολύνει την ανάπτυξη μια βιώσιμη αλληλευτική πολιτική, υπεύθυνη όσον αφορά του αλληλευτικού πόρου, στη δημοκρατία του πράσινου ακροτηρίου και αυτό προ το συμφέρον και των δύο μερών. Το χρηματικό ε, αντίτιμο ε, θα είναι ένα ποσό το οποίο περιλαμβάνει δύο ε, κομμάτια. Το ένα θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόσθετο συμπληρωματικό κονδύλιο θα καταβληθεί από τους Ευρωπαίους που ψαρεύουν στα, κοντά στα νερά του Πράσινου Ακροτηρίου. Η χρηματική αντιπαροχή ε, ετησίως είναι 325.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από τους ε, ε εκεί θα είναι 110.000 ευρώ. Μιλάμε για 100 ευρώ ανατόν ελευόμενο τόνο, 65 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 35 ε, από τους παράγοντες του κλάδου. Μιλάμε για 5.000 ε, τόσους ετησίως ε, εγγυημένη πληρωμή. Επίσης εφάπαξ ποσά που παρέχουν οι εφοπλιστές, άδειες θυναλιευτικού γρηγρή 4.375 ευρώ, 3.150 ευρώ ανά παραγαδιάρικο και 450 ευρώ ανά θυναλιευτικό με καλάμι. Όταν η συνολική ποσότητα υπερβεί τους 5.000 τόνους ενισίων, η ετήσια χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται κατά 65 ευρώ ανά τόνο που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 35 ευρώ ανατόνο που καταβάλλονται από τους πλειοκτήτες ως συμπληρωματική καταβολή, συμπληρωματικό κονδύλιο. Η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν είναι ικανοποιημένη με το γεγονός ότι το ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του πράσινου ακροτηρίου ισούται με εκείνο που κατεβλήθη στο πλαίσιο της εφαρμογής του προηγούμενου πρωτοκόλλου η Επιτροπή Ανάπτυξη χαιρετίζει επίση το γεγονό ότι το πρωτόκολλο αυτό εισάγει νέε διατάξει, δια των οποίων η καταβολή τη χρηματική αντιπαροχή ε, ε, είναι δυνατόν να διακοπεί σε περίπτωση παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων ή δημοκρατικών αρχών το οποίο δεν μα θέτει προβλήματα, διότι το Πράσινο Κροτήρι είναι μια χώρα αρκετά προηγμένη για το ζήτημα αυτό. Τέλο η Επιτροπή Ανάπτυξη επικρίνει την έλλειψη διαφάνεια εκ μέρου τη Επιτροπή, σε σχέση με την κατάταξη στην οποία προβαίνει το θεσμικό αυτό όργανο εκ των υστέρων επιπτώσεων από ένα εξωτερικό ανάδοχο. Η Επιτροπή σας ε, καλεί την Επιτροπή Αλίας ε, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη συνέψη της συμφωνίας. Ωστόσο, έχουμε συντάξει μερικές συνθήκες Πρώτα απ' όλα διαφάνεια των διαδικασιών για την εξακρίβωση των ποσοτήτων που αλλιεύονται συνολικά. Ίσως θα μπορούσε να μας διαφωτίσει λίγο η Κομισιόν από αυτού του ζητήματος, ώστε αυτή η αλία να είναι σύμφωνη με τα κριτήρια διαδοσιμότητας για το πράσινο κριτήρι. Δεύτερη συνθήκη, μεικτή επιτροπή που προβλέπει το πρωτόκολλο μεριμνά ώστε η αικαιρεότητα του συνολικού μηχανισμού της συμφωνίας ως προς τον έλεγχο ως προς τον έλεγχο της διαφθοράς να είναι της υποψίας. Τρίτη συνθήκη, η Μικτή Επιτροπή πρέπει επίσης να επιδιώξει τη λήψη μέτρων για την πρόθεση και να ενισχυθεί η τοπική απασχόληση και άλλες οικονομικές δραστηριότητες και συμπράξεις στον τομέα της αλίας Τέλος, πρέπει να ενισχύσουμε τη λογοδοσία της τοπικής κυβέρνησης που πρέπει να εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των τοπικών αλλιέων, την ανάπτυξη της ε, βιώσιμης βιοτεχνικής αλλιέας σε τοπικό επίπεδο. Αυτά είναι τα ε, κομμάτια για αυτή τη χώρα που παράγει κατά την άποψή μου τον καλύτερο τόνο του κόσμου. Είναι εξαιρετική ποιότητας. Ε, έχει όλες τις δυνατότητες για εξαγωγή. Αυτή η εκθεσή κατά την άποψή μου, ήταν μια έκθεση που ανέλαβα κατά τύχη. Ουσιαστικά είχα την τύχη να συμμετέχω σε μια συνεδρίαση συντονιστών όπου αυτό το είδος έκθεσης ε, συνήθως ε, δίνεται στην προεδρία της συνεδρίασης και έτσι με αυτόν τον τρόπο έλαβα εγώ κατά τύχη ανέλαβα αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ ωστόσο που με βοηθήσατε τόσο πολύ σε αυτό το εγχείρημα και ελπίζω με τη συμφωνία σας ε, είναι η βασική, το βασικό έργο των βουλευτών να κάνουν εκθέσεις. Ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα έχω μια ερώτηση, αν δεν έχει πρόβλημα από αυτού, σε σχέση με αυτή την υπόθεση της αλίας της ε, αλίας Φάλαινα είπε, αλλά δεν είναι φάλαινα, είναι τόνο. Ε, μιλώντας για αυτή τη συμφωνία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον τόνο, αυτό το ψάρι που γίνεται όλο και πιο σπάνιο και ότι ίσως πρέπει να προσέχουμε και ρωτάω λίγο αφελώς. Διαβάζω άρθρα που λένε ότι δεν υπάρχει πια τόνος και ότι δεν πρέπει να ψαρεύουμε άλλο. πολλά ψάρια βέβαια, υπάρχει έλλειψη σε πολλά ψάρια, αλλά ειδικά ε, για τον τόνο διαβάζω και θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορούμε να το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη συμφωνία. Eh, πρώτα πρώτα, συγχαρητήρια στον κύριο Γκέρας για την εκθεσή του, αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε και για την προηγούμενη εκθέση όσον αφορά τον προπολογισμό του 2012. Έχουμε ίδιο συντονιστή μα αλλά τα αλλά και εγώ θα σας συγχαρώ. Οπότε έχουμε αυτό το σχέδιο έκθεση. Θέλω να σας πω τρία πράγματα. Πρώτα πρώτα, νομίζω ότι η ανανέωση του πρωτοκόλου για το πράσινο ακροτήριο μπορεί να βοηθήσει την αληθινή μας πολιτική, αλλά μπορεί να βοηθήσει και το πράσινο κροτήριο για μια πιο βιώσιμη πολιτική, για προστασία των ελληνικών πόρων. Είμαστε πιο υπεύθυνοι στην επιτροπή μας. Ε, οπότε παρακαλώ να λάβει στα σοβαρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα οποία λέμε στην Επιτροπή Αράπτυξη. Έτσι θα βοηθήσουμε την τοπική αιλία. Τέλος, επίσης, έτσι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια σχέση με τι χώρες. Γι' αυτό και Νομίζω θα έπρεπε να μας διευκολύνει η Ένωση, η Επιτροπή, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε όλα τα έργα που χρειαζόμαστε και επομένως να μπορούμε να μας δώσουμε τις Και τώρα. Ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή όσον αφορά την Επιτροπή της Πολιτικής Με λίγες φράσεις να σας παρουσιάσω την συνελευθεία αυτή συμφωνία. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που συνήθει αυτή η συμφωνία. Πρόκειται για συμφωνία, λέγω, που αφορά χώρα, που επαξίως είναι εταίρος μας. Επόμενο στη γενική μας διεύθυνση μπορούμε να πούμε ότι το να ασχολούμαστε με τη χώρα αυτή αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Συμφωνία σχετικά απλή, σχετικά εύκολη, ακριβώ όπω πάρα πολύ σωστά τα είπε ο κύριο Γκέρεν. Ο κλάδος δεν έχει μεγάλες διαστάσεις. Οπότε όλα αυτά τα μυστηριώδη τη σκάφη, ε, το παραγάδι επιφανίας κλπ. Είναι αυτή ελευθερία στερεότητα που δεν απειλεί τις ποσοστώσεις της χώρας. Φυσικά και γίνεται ελέγχη από την ΕΚΑΤ Ο τόνος, ξέρετε, είναι ένα ψάρι. Δεν το ελέγχει μόνο η χώρα. Το ελέγχουν και ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ΚΑΤ. ασχολείται πάρα πολύ με τον έλεγχο αυτό. Επομένω, θεωρούμε ότι η ΚΑΤ είναι ένας οργανισμός που έχει εύρεθμη λειτουργία. Τώρα για να σας πω κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα που ο κ. Γκέρινς μας ε, μίλησε για τον υπολογισμό ε, του συνολικού ελεύματος. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά ε, την αλληλεία. Επομένως υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ υπολογισμού και πραγματικού αλλιεύματος. Προσπαθούμε βέβαια να δουλέψουμε μακρόπνο, να κάνει κάτι και η σχετική χώρα και οι αρχές που έχουμε υπόψη ότι το τι γίνεται με τη διαχείριση, τι γίνεται με τους αλληλευτικούς πόρους, θέλουμε να είναι βιώσιμη αλληλεία. Επίσης, το πλεόνασμα είναι κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί, δεν είναι δυνατόν να αλλιεύουμε ε, κάτι το οποίο δεν αλλιεύει η σχετική χώρα. Αν έλεγε λοιπόν ότι 100% θα αλλιεύει τον τόνο η, χώρα αυτή, θα λέγαμε τόσο καλύτερο θα υπάρχει τότε πλεόνασμα πλεόνασμα είναι κάτι που σχετίζεται με την κατάσταση των ελληνικών πόρων. Είπαμε 100% πλεόνασμα, αυτό σημαίνει ότι είναι σε κάτι κατασκευαστή πόρη και αντίστροφα. Επομένω, κάτι άλλο. Τα περισσότερα ελευτικά στα ανοιχτά. Προδοσιακή αλληλή, δύσκολο να του υπολογίσουμε. Ε, Όντω κάποιοι τοπικοί από το Πράσινο Κροτήριο απασχολούνται στα ευρωπαϊκά σκάφη. Αλλά τέλος πάντων οι πλειοκτήτε στρέφονται σε άλλα κράτη τη περιοχή. Επομένω, έχουμε αυτές τις δύο πτυχές του πρωτοκόλλου για τελείω διαφορετικές. Από τη μία μεριά την εμπορική δραστηριότητα, οι τις δραστηριότητες που για άλλη μια φορά αναφέρω ότι κάτι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλησιώνουν αυτές τις προσπάθειες, άρα είναι το θέμα της παρακολουθής μας και από την άλλη μεριά είναι η τομιακή υποστήριξη που ανταποκρίνει στην ρευτική ε, πολιτική της χώρας, αλλά δεν αντιστοιχεί άμεσα με τον τόνο. Επομένως, έχουμε στη χώρα κάποιους στήματα ελέγχου Και ξέρετε ότι και εμείς ασχολούμεθα και οι έλεγχοι βέβαια χρειάζονται λιγότερο από τις άλλες χώρες της περιοχής. Και δεν κάνουν αυτό που πρέπει όπως η Γουινέα Μπισάου. να βρω τώρα τις ευθύνες των, των, των τοπικών αρχών ή των, τοπικών κυβερνήσεων έχουμε όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε 15 συμφωνίες σχετικές ακόμα και με την Γερλανδία. Γίνεται και διάλογος με τις τοπικές αρχές. Δεν υπάρχουν ναι, ουσιαστικά λάθη. Ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε φυσικά ε, την ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά είναι έτσι γενική ρήτρα που ουσιαστικά δεν αφορά το προσωπικό Όπως είπατε, αφορά άλλες χώρες. Επομένως, πώς θα βοηθήσουμε τις αριθμικές δυνατότητες της χώρας. Αυτό αφορά κυρίως την υπάρχει αλληλεία. Του δοσιακούς αλληλείς. τέλειες διαφορετική δραστηριότητα από αυτή του δικού μας τόλου. Τώρα, όσον αφορά κυρίως διοικητικό πρόβλημα, η πρόσβαση στα έγγραφα, είναι το τελευταίο σημείο, και είναι πρόβλημα αυτό, Κοινοβουλίου και Επιτροπή πρόβλημα το οποίο όμως αφορά μόνο ένα τύπο εγγράφου της ε, μελέτης αξιολόγησης. Όταν μιλούμε για διαφάνεια, για αγαστές ε, ε, σχέσεις θεσμικές, θεσμικών οργανών, εμείς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και καλούμε σε μια τεχνική, τεχνοκρατική συνάντηση το Κοινοβούλιο για διαπραγματεύσεις. Υπάρχει διαφάνεια 100% όσον αφορά τα πρακτικά, όσον αφορά επιτροπές. Βέβαια και υπάρχει διαφάνεια πρόσβαση σε όλα τα νομικά κείμενα. Εμεί μεγάλη μα ικανοποίηση βλέπουμε να ενδιαφέρει τόσο πολύ το κοινοβούλιο και θέλει να συμμετάσχει στις ε, τεχνικέ συνδυάσει. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε συναντήσει που κατατάσσονται έτσι, ούτω ώστε ε, δεν είναι χθε. στις είπαμε θέλουμε να δούμε αφού εγγονίσουμε τη στρατηγική θα πρόκειται για καταιγισμό ιδεών, αξιόλογο. Σε κάποιο πράγμα να συμφωνήσουμε. Γι' αυτό πολλές φορές κατηγορούμαστε χωρίς να ισχύει. Και αυτές οι μελέτες αξιολόγησης περιέχουν πληροφορίες πολιτικά δύσκολες, ευαίσθητε και εμπορικά για τις σχέσεις με την τρίτη χώρα. Γι' αυτό το πράσινο κροτήριο, κάποια στοιχεία όσον αφορά το τζίρο αυτών των πλειοκτητών. Κάποια στοιχεία που στους συμβούλους τα αποκαλύπτουν οι χώρες αλλά δεν είναι δημοσιεύσιμα αναγκαστικά. Όλα αυτά τα οποία έχουν σημασία για τις Οπότε και σε αυτά τα σημεία σημασία θα πρέπει να συζητιούνται. Επομένως, έχουν περιορισμένη σύνθεση συνεδριάσεις. Πολλές φορές. Καταλαβαίνω ότι σα είναι δυσάρεστο, αλλά δυστυχώ αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπετε. Πάντως, μπορείτε όποτε θέλετε να έρχεστε στη Γενική Γραμματεία και να διαβάζετε, μελετάτε μέσα σε περιβάλλον ε, ασφαλές ό,τι θέλετε. Όχι, όχι, ε, εντάξει, δεν μου αρέσει και εγώ να είμαι σε, ένα επόμενο δωμάτιο, αλλά πάντα υπάρχει δυνατότητα. Τώρα και κάτι άλλο, και εδώ θα κλείσω. Αυτές οι μελέτες αποχαρακτηρίστηκαν. Άρα 100% μπορεί να το πείτε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στη γραμματεία της Επιτροπής. Αν θέλετε λοιπόν μπορείτε να έρθετε σε επαφή με αυτούς. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Λοιπόν, ο κύριος Γκέρενς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η απάντηση της Επιτροπής ε, έληξε, έ, ε, εθεσε τέλος αυτή τη συζήτηση και ήταν χρήσιμη διότι για έναν Ευρωβουλευτή είναι δύσκολο να δεχθούμε την ε, περιορισμένη διαδικασία αλλά αντιλαμβάνουμε τους λόγους σας και στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατόν να προβλέψουμε κάποια δυνατότητα να παρακολουθήσουμε εκτάκτως, δηλαδή να μην αποκρύπτουμε τις ε, πληροφορίες, αλλά αν κατάλαβα καλά πρέπει να ακολουθήσουμε τις ενδείξεις ε, της ε, γραμματείας. Εγώ δεν θα καταφύγω σε αυτή την την μέθοδο αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έτσι υπάρχει μία ε, σκοπιμό τη να απομονωθούμε. Ε, και ξέρετε, λέει ο πρόεδρος, και εγώ έχω τα όρια μου. Ε, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι αν πάτε και απομονωθείτε θα μπορέσετε μετά να μας ψιθυρίσατε τι μάθατε. Η κυρία Κέλλερ. Με συγχωρείτε, δεν παρακολούθησα τη συζήτησή σας, αλλά εάν έχουν τη συνήθη φύτους δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Έχουμε μεν ε, ε, πρόσβαση εις ε, το κρυφό αναγνωστήριο, μπορείτε να καθίσετε εκεί που την ε, ε, εποπτεία ενός ε, υπαλλήλου ο οποίος σας παρακολουθεί, δεν μπορείτε να πάρετε αντίγραφα και στη συνέχεια πρέπει να γνωμοδοτήσετε βάσει αυτής της αξιολόγησης των επιπτώσεων την οποία διαβάσετε. Είναι χοντρά και ε, ε, εκτενή έγγραφα και ε, από την άλλη πλευρά έρχεστε και λέτε ναι υπάρχουν προσόντα αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω. Πώς λοιπόν μπορούμε έτσι να συζητήσουμε θέματα που τα θεωρούμε σημαντικά. Νομίζω ότι είναι ένα εμπόδιο. Το συζητάμε ήδη αρκετό καιρό. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν διότι ε, τα έγγραφα αυτά κάποτε ήταν διαθέσιμα. Βέβαια, αν δεν μπορεί κανείς να πάρει σημειώσεις, ε, ξεκινάνε τα προβλήματα. Θέλει να απαντήσει με μία μόνο φράση η Επιτροπή, άντε δύο, πολύ σύντομα. αντί αυτές οι ε, μελέτες αξιολόγησης να αποτελέσουν βάση, ε, μην βασιστείτε αποκλειστικά σε αυτά, αλλά μπορείτε να έρθετε στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και να συζητήσουμε αντί να ε, κοιτάξετε αυτές τις πολύ μεροληπτικές μελέτες, πράγμα το οποίο έχω ήδη επισημάνει. Σας ευχαριστώ. Η ε, καταληκτική ημερομηνία είναι 14 Ιουλίου το μεσημέρι για την κατάθεση των τροπολογιών. Με συγχωρούν οι διερμηνείς, αλλά το κείμενο είναι αγγλικό και θα συνεχίσω αγγλικά. Οπότε, Τώρα θα έχουμε μία συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών με